Hello, good morning everybody. Καλό σας απόγευμα. Πρωτού ξεκινήσουμε, να πω ότι το σημείο 25 αναβάλλεται για τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 λέει ο Πρόεδρος. Το σημείο 25 της ημεσίας So now we go to the point 9. Οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 9 για την προστασία των ατόμων για, ε, στα πλαίσια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος ε, Τζαμπάσκι είναι ο εισηγητής και του δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου Уважаеми господин председател, уважаеми принцип Αγαπητοί συνάδελφοι, υπό το δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα και με το άρθρο 16 της συνθήκης πρόκειται για ένα δικαίωμα που έχει εγγραφεί στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και υπό τον κανονισμό 45 του 2009 αυτό ισχύει και για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεδομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων που θα τεθεί εν που ετέθη εν ισχύ στις 25 Μαΐου 2011 είναι απαραίτητος να αναθεωρήσουμε τον 7 69 ε, με και ως Επιτροπή, μάλλον στην Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων, πρέπει να αναθεωρήσουμε επίσης το όριο ηλικίας των 13 ετών που είναι υπερολικά χαμηλό στα πλαίσια αυτά προτείνουμε η ηλικία αυτή να γίνει 16 έτη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η προθεσμία είναι στις, ε, θα είναι 14 Ιουλίου στις 2.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκη. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη. Ο κύριος Φως, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, πρώτα να ευχαριστήσω τον φίλο Τσαμπάσκι για την έκθεσή του, την οποία έχουμε εξετάσει και στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Για μένα πρέπει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον η συνένεση των παιδιών εντός των θεσμών παίζει κάποιον ρόλο διότι δεν έχω την εντύπωση ότι το θεσμικό μας όργανο έχει απολύτως σχέση με παιδιά. Γι' αυτό και θέτω το ερώτημα κατά πόσον τούτο εδώ παίζει ένα ρόλο. Εάν ταχθεί κανείς υπέρ, άλλωστε το είχαμε και στον βασικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, έχουμε δηλαδή την ηλικία των παιδιών, ε, θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει. Εγώ πάντως θεωρώ ότι πρέπει, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα καθήκον της Νομικής Επιτροπής, αλλά να ευθυγραμμίσουμε την ε, οδηγία με τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων, διότι κάποιοι ορισμοί που έχουν ληφθεί από εκείνο τον κανονισμό δεν λαμβάνονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή ακριβώς ταυτόσιμοι. Πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά ώστε εν τέλει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο σύστημα. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν θα είναι δυνατόν, ε, δεν, μάλλον δεν γίνεται με όλα τα άρθρα του ε, βασικού κανονισμού προστασίας δεδομένων. Και σε ό,τι αφορά Ευρωπόλ και Eurojust, συζήτηση την οποία κάναμε και χθε το απόγευμα ή σήμερα το πρωί, δεν θυμούμε, είχαμε συζητήσει για το εάν τα επιχειρησιακά δεδομένα Ευρωπόλ και Eurojust θα πρέπει να διαχωριστούν από το κείμενο αυτό και να μπουν στην μεταρρύθμιση Europol και Eurojust. Η πρόταση οδηγίας αποτελεί μια γενική ρύθμιση, δεν αναφέρεται ειδικά στην θέση των οργανισμών Europol και Eurojust. Πρέπει πάντως να συζητηθεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες και επαναλαμβάνω την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν καλύτερα, να ευθυγραμμιστεί καλύτερα το περιεχόμενο της παρούσης με τον βασικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η κυρία Χάουταλα, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε επίση το πώς διασυνδέεται ο κανονισμός με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, για παράδειγμα του κανονισμού Ευρωπόλ. Έχουμε από την αρχή μια ξεκάθαρη άποψη σχετικά με το ποιο σύνολο κανόνων υπερτερεί, εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Θα ήθελα να ακούσω από τον εισηγητή κάποια άποψη ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Και αυτό βέβαια δεν είναι μονάχα ζήτημα της σχέσης των ρυθμίσεων που προβλέπονται εδώ με την Ευρωπόλ, αλλά και με Eurojust καθώς και με το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα λοιπόν το τι ακριβώς γίνεται εδώ, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη και του ΣΥΤΟΥ και ίσως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Okay, thank you to everybody. Ευχαριστώ όλους. Σημειώστε παρακαλώ ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 14, όπως είπε και ο εισηγητής. 14 Ιουλίου του 2017, διευκρινίζει η Πρόεδρος. Πάμε τώρα στο σημείο 14. σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 35-2004 της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την αστική ευθύνη για περιβαλλοντικές ε, ζημιές. Σήμερα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες που υπευλήθησαν στο σχέδιο έκθεσης της εισηγήτριας κυρίας Φεράρα, δηλαδή εμού της ιδία και μου δίνω το λόγο και περνώ στα Ιταλικά. Καλό σας απόγευμα λοιπόν και στα Ιταλικά. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σχετικά με την έκθεση αυτή εφαρμογής της οδηγίας της περιβαλλοντικής. Εγώ εξέτασα και έλαβα υπόψη μου τις τροπολογίες σας, τις θεωρώ βελτιωτικές ε, στο κείμενο όχι μόνο βελτιωτικές για την έκθεση, αλλά βελτιωτικές για ένα φάκελο που είναι πάρα πολύ σημαντικός για τους πολίτες, οι οποίοι υφίστανται τις άμεσες συνέπειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το, πρώτο επί του οποίου μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας είναι ότι η βασική κατεύθυνση της εκθέσεως που υπέβαλα εδώ στην Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων παραμένει ανέπαφη. Αυτό με ικανοποιεί. Σημειώνω επίσης ότι ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας όλοι σημείωσαν όχι μόνο τον ανομοιογενή χαρακτήρα της εφαρμογής της αλλά την ανάγκη της ε, καλύτερης, του καλύτερου ορισμού και των κατοφλίων της οποιασδήποτε επίπτωσης ή αντικτύπου περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ε, κύριοι Μπούντα και Τζαμπάσκι δεν συμφωνούν μαζί μου στην επέκταση του πεδίου εφαρμογή ε, της οδηγίας και στις ε, ηλεκτρομαγνητικές ε, επιπτώσεις και τις επιπτώσεις για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ούτε για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις αποζημιώσεις από τις ζημιές που καθορίζει η οδηγία και υποτείνει αυτή, ελπίζοντας και σε μεταξύταση από πλευράς τους, λέω ότι το, ένα τέτοιο ταμείο θα έπρεπε να λειτουργεί υπέρ του περιβάλλοντος και υπέρ των πολιτών σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας και στην οποία περίπτωση θα παρενέβαιναν τα εγγυητικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχω όμως κάποιες απορίες ε, ε, σχετικά με την, ε, τις προτάσεις της κυρίας Χάουταλα σχετικά με την επικυρική ευθύνη του κράτους. Δεν θα ήθελα δηλαδή να σημαίνει αυτό ότι θα το πρόσθετο άκθος της ευθύνη θα το έχουν οι επαγγελματίες πέραν των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να φορτωθούν και το οικονομικό κόστος της οποιασδήποτε αποζημίωσης. Εκτίμησα τις τροπολογίες ε, ε, του κυρίου Γκούτιλαντ σχετικά με την οποιαδήποτε ατμοσφαιρική ρήπανση των οχημάτων που απορρέει από την οδηγία που διέπει τις ε, εκπομπές των οχημάτων όπως και η δημιουργία δημοσίων τραπεζών δεδομένων που θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς που θα διέπεται από την οδηγία. Επίσης, οι τροπολογίες Χρυσόγονου και Μαστάλκα που υπογραμμίζουν τη σημασία δημοσίευσης κάθε περίπτωσης ε, αποδεδειγμένης ε, ευθύνης ώστε να είναι διαφανές και γνωστό σε όλους το κόστος της περιβαλλοντικής ε, αντιστάθμισης. Όλοι επίσης από ό,τι φαίνεται σημειώνουν το, την επίγουσα ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας και προτείνω στους κοιόδης ως εκ τούτου μία και μόνη σύντομη συνάντηση ώστε να συμφωνήσουμε επί κάποιων συμβαστικών τροπολογιών. Αν συμφωνείτε θα μπορούσαμε αυτή τη συνάντηση να την κάνουμε ή στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας και για την πολύτιμη συνεργασία σας. Περιμένω τις απόψεις σας σχετικώς. Ο κύριος Φως έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω να σας μεταφέρω το μήνυμα του σκιώδου συγητού μας κυρίου Ράντεφ, αφού συγχαρώ πρώτα την κυρία Φεράρα για την έκθεσή της. Όλοι βεβαίω θέλουμε να εγγυηθούμε η υψηλά επίπεδα προστασίας της υγείας των πολιτών καθώς και των περιβαλλοντικών προτύπων. Όντως σε πολλές χώρες μέλη σημειώνονται δυσκολίες ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη και ιδίω για την αποζημίωση ζημιών στο περιβάλλον. Πρέπει οι επαγγελματίες και ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα ασφαλιών για την αντιμετώπιση ζημιών στο περιβάλλον καθώς και για την αντιμετώπιση παράπλευρων ε, ε, ζημιών από ατυχήματα που συμβαίνουν. Το ίδιο και για περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας. Πιστεύουμε ωστόσο ότι το ζήτημα της ίδρυσης ειδικού ταμείου πρέπει να εξεταστεί περισσότερο, πιο προσεκτικά. Τονίζουμε ακόμη την πρόταση για τη δημιουργία νέων οργάνων με ελεγκτικές εξουσίες υπό την ισχύ της σχετικής οδηγίας για να περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα να ζητούν οικονομικές εγγύησεις από τα μέρη. Αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο επίσης πρέπει να επανεξεταστεί και σας ευχαριστώ για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου. Η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ Πρόεδρε και η εισηγητά. Σας ευχαριστώ για το σχέδιο αυτό εκ μέρους της ομάδας. Πιστεύω ότι το κείμενο αυτό τοποθετείται σε ένα πεδίο πολλών ανησυχών που είχαμε εδώ και χρόνια για την εφαρμογή της οδηγίας. Το πεδίο της εφαρμογής της οδηγίας αυτής ήταν εξαιρετικά περιοριστικό και είχε και κενά. Πρέπει λοιπόν να παράσχουμε έμπνευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει σε μια αναθεώρηση και επανεξέταση της οδηγίας. ως εισηγήτρια δεν είστε απόλυτος υπέρ της προτάσεως αυτής της υποχρεωτικής ευθύνης από πλευράς του κράτους, αλλά πρέπει να δει κανεί πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κατά την οποία έχουμε διαφορετικά πρότυπα και πώς θα πληρώσουμε τα κενά αυτά. Εγώ θα υποστήριζα την ιδέα σας της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου που θα κάλυπτε περιβαλλοντικές ζημιές που δεν καλύπτονται από το ELD ή από κανονικές χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις, δηλαδή φυσικών καταστροφών. Αυτό θα κάλυπτε ένα κενό Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τους ταχαίως τροποποιημένους ε, επιμολυντές τους περιβαλλοντικούς τροποποιούμενους μάλλον. Πρέπει επίσης να καλύψουμε την οποιαδήποτε ζημιά ε, στο οικοσύστημα, δηλαδή στη χλωρίδα και την πανίδα, όπως και να βοηθήσουμε φορείς και ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να χρησιμοποιούν ασφαλιστικά συστήματα ευρύτερα και πιο συχνά σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς. Και ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και την υποχρεωτική κάλυψη των οικονομικών φορέων που δρούν στο πεδίο αυτό, υπό το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Νομίζω 10 τροπολογίες έχουν υποβληθεί στο όνομά μου και απλώς να αναφέρω την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για τους φορείς, την περιβαλλοντική δηλαδή, διαφορο, διαφοροποιημένα κατέφλια μέγιστη ευθύνη, επέκταση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία για να καλύπτει και τη δημόσια υγεία, υποχρεωτική επικουρική αστική ευθύνη του κράτους και παράληψη ε, τον μηχανισμό να μείνει ώστε να προαγάγουμε την αρχή του ότι ο, ο πληρώνει τη ζημιά. Επι, όπως επίσης και μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Ε, περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια καλή ισορροπία μαζί με εσάς και με τους άλλους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Η έγκριση στην ε, Γιούρη είναι για τις 7 Σεπτεμβρίου. Okay, so now we can start with the hearing. Dear speakers, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σε αυτή την ε, δημόσια κρόση για, αυτό, για την διαδικασία υποταστικό δίκαιο που έχουμε διοργανώσει για σήμερα. κανόνες λοιπόν πολιτικής δικονομίας μετά την νομοθετική έκθεση του κύριου Χράντεκ ε, για, τις, ε, για τους κοινού κανόνες της δικονομίας ώστε να εφαρμόζονται τα ουσιαστικά δικαιώματα των υποκειμένων ή στις ε, διαδικασίες τις δικαστικές το οποίο συνδέεται με το θεμελιώδες δικαίωμα σε δίκαιη εξέταση και δίκαιε υποζημιώσει υπό τον, τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων άρθρο 47 όπως και την ε, συνθήκη ε, στο άρθρο 6. Το Μάιο του 2014 εκκίνησε ένα έργο ε, όπου εξέταζε τους περιφερειακούς κανόνες της δικονομίας η Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων και ο κύριος Σβόποντα υπήρξαν θεσμικός παρατηρητής του έργου αυτού και παρακολούθησε στενά την πρόοδό του σε όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Η πρώτη ενοποιημένη εκδοχή στα αγγλικά υπευλήθη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ουνιντρουά στις 11 Μαΐου στη Ρώμη. Η ακρόαση αυτή μετά την παρουσίαση στο Συμβουλίο για την πρόσβαση στα αποδεκτικά στοιχεία όπως και στα μεταβατικά και προστατευτικά μέτρα και εν ώψη των επόμενων βημάτων του έργου αυτού θα διεξαχθεί με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αστικού Δικαίου που υπήρξε και συντονίστρια της ομάδος ALDE και εισηγήτρια για πολύ σημαντικούς φακέλους εδώ στο Κοινοβούλιο όπως και αντιπρόεδρος υπήρξε. Η κυρία Βόλης, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Φεράρα και βεβαίω για τα ευγενικά σας λόγια. Είναι για μένα πάντοτε μεγάλη χαρά να επανέρχομαι στα έδρανα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρισκόταν στην καρδιά των ε, βουλευτικών μου δραστηριοτήτων όταν ήμουν ευρωβουλευτή. Θα ήθελα πρώτα να απευθύνω συγχαρητήρια και στον εισηγητή σα και στην Επιτροπή σα για την τελική έκβαση τη εκθέσεώ σα στο σημαντικό αυτό τομέα. Η έκθεση Ράντεφ από, πολλούς, από πολλές απόψεις είναι συμπληρωματική της εργασίας του Ινστιτούτου μας Ευρωπαϊκού Δικαίου και UNIDROIT και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε για τον τρόπο με τον οποίο η Νομική Επιτροπή και η Γραμματεία σας συνεργαστήκατε πολύ στενά μαζί μας. Αυτό που θα ήθελα να κάνω τώρα, σύντομα δηλαδή, στην παρουσίασή μου, είναι να σας δώσω μια αίσθηση του πού βρίσκεται τώρα η εργασία μας αυτή, να ρίξω φως σε κάποιες από τις διαφορέ ανάμεσα στα όσα κάνουμε εμεί και στην έκθεση που έχετε συντάξει εσείς και τέλος να σας ε, δώσω και μια κατεύθυνση, δηλαδή του πού βρισκόμαστε, προς τα πού κινούμεθα. Είμαι θα ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρακολούθησε προσεκτικά και με κριτικό πνεύμα την εργασία μας και νομίζω ότι και εμείς οι ίδιες αλλά και εσείς με την έκθεσή σας θα πρέπει να το θεωρήσετε αυτό ως καλό σημάδι ότι κάτι θα προκύψει από όλη αυτή τη δραστηριότητα. Ελπίζω να λειτουργήσει το μηχάνημα προβολής των διαφανειών. Όντως, ναι. Βλέπετε λοιπόν ε, ένα σύντομο ιστορικό για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλούμε. Το project Eli Unidroa ξεκινά από μια παλαιότερη εργασία που είχε δημοσιευθεί το 2004 από το American Law Institute και UNIDROIT με στόχο, με, μάλλον με τίτλο «Αρχές υπερεθνικών ε, δικονομικών κανόνων». Αυτό που θέλουμε εμείς τώρα στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δικαίου, Ινστιτούτο Δικαίου και UNIDROIT να θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να φτιάξουμε συγκεκριμένους κανόνες ξεκινώντας από εκείνες τις αρχές διαδικασίας αναγκαστικής που θα επιβάλλεται όμως ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και γι' αυτό το έργο αυτό έχει τόση σημασία και ε, για την δική σας δουλειά. Κατά κάποιο τρόπο η δική σας εργασία σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα είναι εγκύτερα στις αρχές, στις βασικές αρχές από την άποψη του που βρίσκεται. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να δώσουμε το επόμενο λεπτομερέστερο βήμα προβλέποντας συγκεκριμένους δικονομικούς κανόνες που θα ισχύουν για τα δικαστήρια και τους διαδίκους. Ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί το project αυτό είναι βασισμένο στις εργασίες διαφόρων ομάδων εργασίας και κάθε μια από τις ομάδες εργασίας έχει δύο εισηγητές Μία από τις εισηγήτριες αυτές είναι δίπλα μου εδώ στα αριστερά μου με το ροζ που κάμισο και θα σας εξηγήσει τις λεπτομέρειες μιας από τις ομάδες εργασίας μας. Δεν ε, έχουμε στόχο να παραγάγουμε νομοθεσία. Πρόκειται για soft law instrument, για εργαλείο δηλαδή ατελούς ή ήπιου δικαίου. Έχουμε όμως την πολυτέλεια σε κάθε ομάδα εργασίας να ε, συμμετέχουν ε, πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι από τις διάφορες δικαιοδοσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ε, γι' αυτό ε, το έργο μας έχει προχωρήσει και έχει επιταχύνει από το 2014. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και είναι πραγματικά σχεδόν δύσκολο να τους κρατούμε μακριά από τις συναντήσεις μας. Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τη συνεχιζόμενη εργασία μας. Για να σας δώσω μία ιδέα, οι πρώτες τρεις ομάδες εργασίας που έχουν αρχίσει και των οποίων η εργασία τώρα ε, αρχίζει να συνδυάζεται, να συγχωνεύεται, είναι πρόσβαση σε πληροφορίες, προσωρινά και μέτρα και η επίδοση εγγράφων. Εάν δείτε τη δική σας έκθεση, θα δείτε ότι καλύπτεται κάποια από τα θέματα αυτά, τα οποία είναι κέρια για την πολιτική δικονομία, και για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της. Για να σας δώσω τώρα μία αίσθηση για τα ποια θέματα, ποια θέματα μας απασχολούν περισσότερο. Είναι οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που και τα δύο θέλουμε να είναι προοδευτικά με την έννοια ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πράγματα όπως η video conference. Τώρα προσωρινά και μέτρα προστασίας εδώ πρόκειται για μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε κάποιον ο οποίος θέλει να ε, κάνει μια αγωγή, φοβάται όμως ότι μπορεί να εξαφανιστούν τα ε, στοιχεία. Από την άλλη μεριά πρέπει βεβαίως να προστατευτούν και τα δικαιώματα του εναγωμένου και αυτά είναι δύσκολα να εξισορροπηθούν σε οποιαδήποτε ένομη τάξη. Βλέπω όμως να διαφαίνεται και η τάση αυτή και στη δική σας ε, δουλειά. Τέλος η επίδοση των εγγράφων. Εδώ είναι η ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε κάτι το πολύ σύγχρονο με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να επιδίδονται τα έγγραφα ε, με πολύ σύγχρονο τρόπο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι κοινά στο έργο και των δύο πλευρών, και το δικό μας και το δικό σας. Ωστόσο θα δείτε ότι εμείς έχουμε προχωρήσει σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες με τα όσα έχουμε κάνει και σε λίγο θα σας εξηγήσουμε και άλλα πράγματα. Σχετικά με τις άλλες διαδοχικές ομάδες εργασίας που αναφέρονται σε άλλα ε, θέματα πολιτικής δικονομίας, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ προφανή και αυτά που σας γράφω στη διαφάνεια. Εγώ πρόσθεσα στο τέλος, και αυτό είναι και το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο του project, δηλαδή ε, ε, μεγαλώνει διαρκώς και ταχύτατα. Έχουμε άλλη μια ομάδα εργασίας δηλαδή που ε, ε, ασχολείται με τις εφέσεις. Ανακαλύψαμε δηλαδή ολόκληρη την πολιτική διαδικασία, τη διαδικασία ενώπιν του πολιτικού δικαστηρίου. Αυτό που τονίζουμε εδώ και νομίζω έχει ενδιαφέρον αλλά και δυσκολία είναι οι υποχρεώσεις των μερών, των διαδίκων δηλαδή και των δικηγόρων. Πρόκειται για κάτι που θα δείτε, εάν εξετάσετε την εργασία μας, που ε, διαχέεται και μέσα στο έργο όλων των ομάδων εργασία, Δηλαδή, με άλλα λόγια, πώ τα μέρη και οι δικηγόροι θα συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Πάλι όμως δεν είναι και εύκολη υπόθεση να επιδευτεί αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει επίσης είναι ότι και εσείς είδατε στην εργασία σας την σημασία του ρόλου του δικαστού αυτό είναι μια συζήτηση η οποία προκαλεί πολλές δυσχέρειες σε εμά, διότι υπάρχουν διαφορετικές νομικές παραδόσεις και με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι έχετε καταφέρει να το περάσετε το σημαντικό ζήτημα, δηλαδή τον διαχειριστικό ρόλο του δικαστηρίου και του δικαστού στην έκθεσή σας, γιατί καταφέρατε να το συζητήσετε αυτό και εμείς βέβαια το επεξεργαζόμαστε με περισσότερη λεπτομέρεια. Βέβαια, είδα επίσης ότι εσείς ε, προχωρείτε και κάπως περισσότερο ε, σε ό,τι αφορά το εξωτερικό πλαίσιο γύρω από την πολιτική δικονομία ε, με πράγματα όπως δικαστικά τέλη, όπως δικαστική αρρωγή και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Από την άλλη μεριά δεν βρίσκουν θέση στη δική μας δουλειά, της οποίας το αντικείμενο είναι κυρίως η λεπτομέρεια της κίνησης της διαδικασίας. Τώρα που έχουν πάρει μπρος όλες αυτές οι ομάδες εργασίας και όπως είπα οι πρώτες τρεις έχουν ήδη συντάξει ας πούμε ημιτελειοποιημένα σχέδια, θα χρειαστεί να συνδυάσουμε όλη αυτή τη δουλειά. Και για το λόγο αυτό την τελευταία χρονιά δημιουργήσαμε κάτι που το είπαμε δομική ομάδα, structure group, και όπου πραγματικά αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον τη δουλειά, τις οποίες ηγούνται δύο σημαντική πανεπιστημιακή, Σάντρα Κράμερ και Λοίκ Καντέ, ο Λοίκ ο οποίος ε, έχει εμπλακεί και στην εργασία του Ανικού Ινστιτούτου Δικαίου και αυτό που κάνουν τώρα για δικό μας λογαριασμό είναι να ε, φτιάξουν ένα ενίο σύνολο από όλη αυτή προσπάθεια επιβλέποντας και την ουσιαστική αλλά και την γλωσσική ε, προσπάθεια, δηλαδή συντονισμό ουσιαστικό και γλωσσικό. Μπορείτε να φανταστείτε τα προβλήματα που έχετε και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο με τον συντονισμό του έργου διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών γύρω από μια έκθεση, ε, περίπου τα ίδια αντιμετωπίζουμε και εμείς και μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι, ποιος είναι ο βαθμός σχέδιας. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα λειτουργικό σύνολο το οποίο θα διέπεται από κάποια συνοχή. Το τελικό κείμενο θα συνταχθεί σε αγγλικά και γαλλικά ώστε υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν και τα γλωσσικά θέματα. Να πω λίγα λόγια τώρα για την αναφιόμενη δομή, αν μπορώ να την πω έτσι, έχουμε ένα κοινό σχεδιασμό για κανόνες και σχόλια επί αυτών, ένα template δηλαδή, ένα συνεκτικό τρόπο σύνταξης με παρόμοιο αριθμό λεπτομεριών ώστε να διατηρηθεί μια ενιαία μορφή στο κείμενο ώστε να μην είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα των εργασιών των διαφορών ομάδων εργασίας. Όπως είπα, συντάσσονται στα αγγλικά και στα γαλλικά. Η διαρθρωτική ομάδα, η δομική ομάδα, η structure group, έχει λάβει feedback από τις πρώτες τρεις ομάδες εργασίας και αυτό μας βοήθησε να δούμε κάποιες από τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε. Έχει ξεκαθαρίσει το πεδίο εφαρμογής, το scope, θα αναφερόμαστε μόνο σε αστικά και εμπορικά θέματα, όχι γαμικές διαφορές, όχι γονικές παιδιών κλπ. Αρχίζουμε επίσης να βλέπουμε ότι Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία και ε, σε κάποιο βαθμό επικαλύψεις μεταξύ του έργου των διαφόρων ομάδων εργασίας. Είπα ότι πρόκειται για ε, τον τρόπο, για αυτό, για αυτό που βλέπουμε δηλαδή και νομίζω ότι είναι περίπου αναπόφευκτο υπό ορισμένε ε, συνθήκες να προβλέψουμε και εναλλακτικού κανόνες που να σέβονται τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις. Εδώ μπορώ να σας δείξω απλώς ε, ένα ενσταντανέ, μια μικρή φωτογραφία, δεν τα διαβάζετε από μακριά βέβαια αυτά, αλλά κινούμεθα προς την κατεύθυνση σύνταξης ενός κειμένου, ενός εγγράφου, που θα έχει τη μορφή κώδικα, ας το πω έτσι, το λέω έστω και αν είμαι ε, Αγγλίδα ε, που για μας οι κώδικες είναι ε, έχουν κάποια όλο ιδιαίτερη σημασία, αλλά πάντω αυτό ε, θα είναι ε, το, η μορφή. Θέλω να πω τελειώνοντα ότι υπάρχουν προσδοκίες σε ό,τι αφορά ένα συνολικό τελικό σχέδιο κάποια στιγμή περί τα τέλη της ανοίξεως του 2018 και τελικό έγγραφο αρχές του 2019. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προβλέψει και βλέπω από το ψήφισμα που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ και στην ανταπόκριση από μέρους τους. Ελπίζω ότι σας ε, έδωσα μια επαρκή επισκόπηση του που βρισκόμαστε και σας κατέδειξα και την συμπληρωματικότητα του έργου μας ως προς το δικό σας και ελπίζω με κοινή προσπάθεια να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα της πολιτικής οικονομίας είτε είναι μέσα στην Ευρώπη η πατρίδα μου είτε όχι, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Σας ευχαριστώ κύριε Γόλης για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Τόσκρουπ έχει το λόγο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα και συνεισηγητής της ε, ομάδας εργασίας. Three working groups. So please, Dr. Torsgroup, you have the floor for 15 minutes. Για θέματα επίδοσης εγγράφων έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμότατα την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την πρόσκλησή της. Είναι τιμή για μένα το ότι εκπροσωπώ το πρόγραμμά μας μαζί με την κυρία Wallace, μέλο της ομάδας για το διατύπωση του τελικού εγγράφου. Ξεκίνησε το 2014 η προσπάθεια και εγώ ασχολούμαι ειδικότερα με το θέμα της επίδοσης νομικών εγγράφων μαζί, με τον καθηγητή Στάντλερ από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας. Να σας δείξω λίγο το, τη σύνθεση της ομάδας. Στις υπόλοιπες ομάδες εργασίας είναι η Wendy Κένετ από το Cardiff, ο κύριος Τσικρίκας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κριστόφορο από την Πάντοβα, και ο Εμμανουέλ Ζελόν από το, Παρίσι 1 Πανθέων Σορβόνη. Ο κύριος Κριστόφορο και εγώ ασχολούμεθα και με την δικηγορία. Ξεκινήσαμε το 2014 και μετά από δυόμιση χρόνια δουλειάς το 2014 ε, είχαμε 16 συγγνώμη, ολοκληρώσαμε το βασικό κομμάτι της δουλειάς μας. Όπως είπε η Diane Wallace, αυτές οι τρεις πρώτες ομάδες εργασίας έχουν υποβάλει πλέον τα, τις τελικές τους σχεδόν διατυπώσεις και θα ενσωματωθούν στο τελικό έγγραφο ή έχουν μάλλον ενσωματωθεί και παρουσιάστηκαν τον μήνα Μάιο στο Συμβούλιο το Διοικητικό. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και τη διαφορετική ομάδα η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πιο συστηματικά. Συνεργαζόμαστε και με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης που ασχολείται με το θέμα του κόστους. Και τώρα ξεκίνησε η εργασία της συγκεκριμένης ομάδας will only not have time to deal with, with all these uh, three parts of... Λοιπόν, ε, υπάρχουν τρία τμήματα κανόνων. Δεν είναι τόσο λεπτομερής όσο οι ε, εθνικές δικονομικές ρυθμίσεις, αλλά παρόλα αυτά Νομίζω ότι έχετε μία πρώτη διατύπωση ε, ε, η οποία είναι παράρτημα στην ανάλυση η οποία είχε αποσταλεί τον Ιανουάριο του 2017. Θα αναφερθώ σε ε, τρεις ομάδες της εργασίας της ομάδας επιδόσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικές θα μιλήσω για τους ε, στόχους, θα μιλήσω για την ηλεκτρονική επίδοση και θα μιλήσω επίσης και για τον συσχετισμό των επιδόσεων με άλλους τομείς και τελικά για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αν έχω χρόνο μετά από αυτά, ε, θα αναφερθώ πολύ σύντομα και σε κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις τις οποίες έχω να κάνω σχετικά με την έκθεση Ράντεφ. Αυτό δεν εκπροσωπεί βέβαια την ομάδα της, του, στο σύνολο της ομάδας, αλλά μόνο την δική μου προσωπική άποψη ως πανεπιστημιακού ερευνητή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην διαδικασία δουλειάς. Οι διάφοροι πανεπιστημιακοί έχουν εκπλαγεί από το ιδιαίτερα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και οι συνάδελφοι στο UNIDROIT οι οποίοι έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν κανόνες και να εξυγχρονίζουν νομικές ρυθμίσεις μας είπαν ότι ο χρόνος είναι αρκετός. Αλλά έχουν υπάρξει πάρα πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα και για το ίδιο το χρονοδιάγραμμα. Ε, χρειάστηκαν δυόμιση χρόνια ε, στην πρώτη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε χρόνο να σκεφτούμε, να χωνέψουμε σε εισαγωγικά τις απόψεις των άλλων ομάδων, τους δίδαμε ε, κανόνες και στις υπόλοιπες ομάδες και στην ε, Διοικητική Επιτροπή και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Ρόσλερ, και στον παρατηρητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων κοινοτικών οργάνων. Οργανώσαμε επίσης και μια μεγάλη δημόσια εκδήλωση και μπορέσαμε να προχωρήσουμε σε βάθος, να αναθεωρήσουμε και να οδηγηθούμε σε ένα προϊόν στο οποίο εμείς έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει λοιπόν εδώ μέσα στη δουλειά που έχουμε κάνει μια υψηλή δόση υπομονής για να έχουμε ένα τελικό προϊόν ουσιαστικό το οποίο να συνοδεύεται από ένα φιλόδοξο συνολικά χρονοδιάγραμμα. Τώρα, ε, σε σχέση με το πρώτο τμήμα, στην ομάδα επιδόσεων, εμείς είπαμε ότι διαπιστώνουμε την ύπαρξη διαφορετικών κανόνων διασυνοριακών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι για τις εσωτερικές διαδικασίες. Καταλήξαμε λοιπόν σε κάποιους γενικούς κανόνες που μπορεί να εφαρμόζονται και στις διασυνοριακές και στις αυστηρά εσωτερικές εθνικές ρυθμίσεις. Στην ουσία δηλαδή μετακινήσαμε το τέρμα προς τα εμπρός, κάναμε ένα άλμα από τη συζήτηση η οποία γίνεται στην Ευρώπη σήμερα, έτσι ώστε οι επιδόσεις να είναι παρόμοιες και σε εσωτερικό επίπεδο και σε επίπεδο διασενοριακό δεν απαιτείται να υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό παράλληλο σύστημα και παράλληλοι κανόνες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι επιπλέον κανόνες για τις διασυνοριακές ρυθμίσεις ε, για θέματα όπως η μετάφραση. Και τώρα περνάω στο δεύτερο, αν θέλετε, ε, θέμα, είναι η ηλεκτρονική επίδοση. Ε, είναι κάτι το οποίο από τη φύση του αν θέλετε ξεπερνάει τα σύνορα. Εγώ μπορώ να είμαι στην ΚΟΑ και να μου επιδοθεί ένα, ε, ένα έγγραφο μέσω του επαγγελματικού μου email. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο στην ουσία εξαφανίζει τα σύνορα και είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει και σε ε, διαφορετικά επίπεδα το σενάριο της ηλεκτρονικής επίδοσης. Ε, θέλει κανείς να επιδώσει μια υποχρέωση σαν παράδειγμα σε πολίτες ή σε άλλα νομικά πρόσωπα καταγραφής και διαθεσιμότητας αποδοχής επιδόσεων και πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ τίθενται σοβαρά θέματα ελευθερίας και ιδιωτικότητας και σημαντικά θέματα για την σχέση κράτους-πολίτη και ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και τον πολίτη τον μεμονωμένο από την άλλη. Προσπαθήσαμε εμείς να υπογραμμίσουμε διαφορετικά ηλεκτρονικά μέσα επίδοσης το κάναμε με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές μορφές επίδοσης. Υπογραμμίσαμε εμείς την τελική μας πρόταση, στο τελικό μας προϊόν, ότι απαιτείται να υπάρχει επιβεβαίωση, απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, ανεξάρτητα από τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιούμε. Στα πλαίσια της μεθόδου αυτής συμπεριλάβαμε σαν παράδειγμα και τα ηλεκτρονικά μέσα. Συμπεριλάβαμε τα ηλεκτρονικά μέσα και ε, την περίπτωση αγνώστου διαμονής πολιτών ή και κάποιες άλλες μεθόδους ε, τελευταίας τελικής προσφυγής θα έλεγα για να μπορέσουμε να επιδώσουμε. Υπάρχει επίσης και συμπερίληψη ενός ε, σημαντικού ε, θέματος, ε, μια σημαντικής αν θέλετε ρύθμισης που αφορά το Συμβούλιο σχετικά με τη διαθεσιμότητά του να αποδέχεται έγγραφα κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεώς του και ταυτόχρονα όταν αλλάζουν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τίθεται η υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι μια διαδικασία θα έλεγα ε, σχετικά ε, αδιάκριτη. Από την άλλη ε, εξαρτάται, εξαρτάται από το τι επικρατεί στη συγκεκριμένη χώρα και από το ποιοι είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές αν θέλετε. Δηλαδή είναι οι περιφερειακοί εταίροι αυτοί που έχουν την ευθύνη. Είναι οι διάδικοι ή το δικαστήριο που είναι αρμόδιοι και έχουν προτεραιότητα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να συνειδητοποιήσει κανείς ότι οι κανόνες για την επίδοση δεν είναι νομικές ρυθμίσεις, αλλά βρίσκονται σε διαδραστική σχέση με άλλες ομάδες εργασίας στο συνολικό πρόγραμμα. Οι ομάδες αυτές επίδοσης, η ομάδα επίδοσης συνδέονται επίσης και με αυτό το οποίο είπε η Νταϊάννα ε, ποιοι άλλοι είναι οι εταίροι, είναι κλητήρε, είναι ιδιώτες κλητήρες, είναι κλητήρες κρατικοί του δημοσίου. Ε, εμείς δεν ασχολούμαστε με το θέμα αυτό παρά μόνο περιφερειακά, αλλά σε εσωτερικό επίπεδο ιδιαίτερα είναι σημαντικό να κατανοήσει ότι ε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς βλέπει κανείς το πρότυπό μας, το μοντέλο μας και πώς μπορεί είτε να απομονωθεί από αυτό είτε να συσχετιστεί με αυτό. Συνεπώς λοιπόν είχαμε, δείξαμε κάποιο πραγματισμό, είπαμε ότι οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι διασυνοριακής φύσεως. Εδώ ίσως στήθεται και ένα θέμα, αν θέλετε συμπεριλάβαμε και κατά κάποιο τρόπο ένα τμήμα της επικουρικότητας στο σχέδιό μας. Να πω επίσης και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό εμείς όταν συζητάμε τα θέματα αυτά το κάνουμε και στα πλαίσια των διαφορετικών ομάδων εργασίας και στα πλαίσια των γενικότερων συναντήσεων και το σχέδιό μας δεν έχει σχέση να βρούμε μια κατελάχιστον κοινή λύση σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Υπάρχει μια εύκολη τάση θα έλεγα όπως είπε και ο Άντερς ε, να ενιοποιούμε προς τα κάτω, μόνο και μόνο για να βρούμε έστω ένα ελάχιστο κοινό χώρο. Ενώ αντίθετα ε, η δική μου ομάδα εργασίας προσπάθησε να ε, προτείνει ένα μοντέλο, ένα πρότυπο το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι ξεπερνά την ελάχιστη κοινή λύση του τι ισχύει δηλαδή σήμερα σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρώπη. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στις εγκάρσεις μορφές συσχετισμού της δικής σας έκθεσης και της δικής μας εργασίας. Εγώ διάβασα την έκθεσή σας, παρακολουθώ από κοντά τις εργασίες σας τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και το ενδιαφέρον σας για τις αστικές διαδικασίες. Ε, υπογραμμίζω την ποιότητα της δουλειά σας και θεωρώ ότι είναι σημαντική. Όμως, σε επίπεδο soft low, θα μπορούσε κανείς να πει ότι για να υποστηριχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί επιπλέον αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συνεργαζόμενους στον τομέα το νομικό στην Ευρώπη, πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Ποιος αναλαμβάνει δράση, πού και πώς. Και όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό έχουν διαφορετικές ίσως απόψεις. Οι πανεπιστημιακοί που ασχολούνται με τις αστικές διαδικασίες θεωρούν ότι θα πρέπει να θέτουμε κάποιους στόχους με, τριόφ, με να κάνουμε προτάσεις και να αφήσουμε ε, όργανα όπως ε, το δικό σας και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να το κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι επιθυμούν με αυτό και να αλληλοεπιδράσουν ίσως με τις προτάσεις των πανεπιστημιακών. Πάντως, μια διαδικασία εκ των άνω δεν είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι η προσθήκη νέων στρωμάτων διαδικασίας, νέων σταδίων διαδικασίας είναι κάτι το οποίο δημιουργεί θέματα και στους νομοθέτες σε εθνικό επίπεδο. Αν ενδιαφερθούν όμως αυτοί στο δικό μας μοντέλο, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ευρύτερο θα έλεγα μοντέλο, μια ευρύτερη προοπτική και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Θα περάσουμε στο τρίτο τμήμα τώρα. ο αρμόδιος για νομοθετικά θέματα στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε να μας παρουσιάσει την πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα. Έχει το λόγο κύριε Ρώσνερ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα ή μάλλον καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Με, να με συμπαθάτε που ήρθαμε κάποια καθυστέρηση. Ε, τα τρένα καμιά φορά καθυστερούν. Ε, λυπούμε που δεν άκουσα την ε, παρέμβαση της κυρίας Γουάλης που είμαι βέβαιος ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον και σας έδωσε η Γενική Επισκόπηση του έργου. Εμείς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε παρατηρητές. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του project με μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αποτελεί καλή ιδέα η οργάνωση μιας δημόσιας ακρόαση για το θέμα αυτό και πιο συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο project. Πρώτα λοιπόν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία οργάνωση δημόσια ακρόαση για το σημαντικό θέμα. Να αρχίσω δίνοντα συγχαρητήρια και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου και στο UNIDROIT, στο Διεθνές ε, ε, Ίδρυμα Ενοποίησης του Αστικού Δικαίου για την τελικοποίηση του έργου σχετικά με την επίδοση εγγράφων, την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και στα προσωρινά και μέτρα ασφάλεια ή ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπερβάλλω εάν πω ότι εξετάζουμε και την έκθεση Storm γιατί είναι σαν σημείο αναφοράς και ταυτόχρονα θα εξετάσουμε και την έκβαση των Ιδρυμάτων ELI και Μητρουά για πολλά χρόνια ως πραγματικά state το the σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα του δικαίου. Παρακολουθούμε την εργασία αυτή με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται να συμβάλλουμε με σχόλια, παρατηρήσεις σε διάφορες ε, περιπτώσεις, σε διάφορες ευκαιρίες και βεβαίως μια φορά δίνεται και συνέχεια στις συστάσει μας. Θεωρούμε ότι το έργο που εκτελούν τα δύο ιδρύματα είναι και μια πολύτιμη ε, πηγή έμπνευση που μπορεί να συμβάλλει και στον περαιτέρω προβληματισμό για την προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θεσπίσει και στον τομέα αυτό η συνθήκη. Από τη δική μας οπτική υπάρχουν τρεις, τρία σημεία της ε, αστικής εν προκειμένου της πολιτικής οικονομίας, δηλαδή αφενός η αναγνώριση των αποφάσεων. Δεύτερο, αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία σε ζητήματα αστικού δικαίου. Τρίτο, η οπτική των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και οι τρεις αυτές οπτικές γωνίες ε, διασυνδέονται μεταξύ τους και το δικονομικό δίκαιο έχει βεβαίω ε, ε, επηρεάζει και τις τρεις αυτές πτυχές. Να εξηγήσω. Δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στο περιφερειακό επίπεδο χωρίς αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και δεν μπορεί να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη χωρίς σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβαση στην δικαιοσύνη και το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνουν και το δικαίωμα σε μια αποτελεσματική και ταχεία πολιτική δίκη. Διότι καθυστέρηση στην ε, απονομή δικαιοσύνη σημαίνει στην ουσία άρνηση δικία. Διότι στερείται, στερείται περιεχομένου η δικαιοσύνη εάν καθυστερεί υπερβολικά το δικαστήριο ή αν ε, δεν μπορεί να γίνει εκτελεστή η απόφαση. Η πολιτική δικονομία προβλέπει τις αναγκαίες ε, προστασίες και διευκολύνει την ομαλή κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων, εγγυόμενη έτσι και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα στοιχεία που διέπουν την ε, σκέψη μας όταν συμμετέχουμε στο έργο αυτό. Είμαστε δε πεπισμένοι ότι τα μέλη των διαφόρων ομάδων εργασίας συμφωνούν με τους στόχους αυτούς. Ως παράδειγμα, όπως εξήγησε μόλις η Εύα, η νέα προσέγγιση για το έργο που γίνεται από την ομάδα εργασίας επίδοσης της ε, εγγράφων, ξεκινώντας από τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις για να καταλήξουν σε ένα ενιαίο κεφάλαιο που θα καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις, βέβαια με κάποιους ειδικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται σε διαμεθοριακές ε, υποθέσεις για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις μεταφράσεις δείχνουν ότι τα στοιχεία που έχουν ε, σημειωθεί λαμβάνονται υπόψη στην εργασία αυτή και θεωρείται ότι η εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελεί μέσον για την αύξηση της εμπιστοσύνης γενικότερα αλλά και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πιο συγκεκριμένα ώστε εν τέλει να προωθείται η αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτού του είδους η προσέγγιση και πάντως αυτή η στάση ε, γίνεται δεκτή από πολλές ομάδες εργασίας. Αναγνωρίζω το γεγονός ότι ο βασικός στόχος του έργου το project δηλαδή, είναι η εθνική νομοθεσία, δηλαδή να φτάσει μέχρι την εθνική νομοθεσία. Ναι. Βέβαια, η πολιτική δικονομία που λειτουργεί στο εθνικό επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί ή να βελτιώσει τις διαμεθοριακές νομικές σχέσεις ό,τι αφορά την επίδοση των δικογράφων, την ε, πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία και εν τέλει πάλι να δημιουργήσει ένα πραγματικό χώρο απονομής δικαιοσύνης όπου διακινούνται ελεύθερα οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν είμαι εκ των βασικών αγοριτών και γι' αυτό θα αρκεστώ σε αυτά τα λόγια για την ώρα που απλώς συμμετέχω. Θεωρώ ότι το έργο είναι σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής δικονομίας και είμαστε πεπισμένοι ότι η τελική έκβαση θα συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη του σημαντικού αυτού τομέως του δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρος κυρία Φεράρα, ευχαριστώ κύριε Ρόσνιλ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ποιος θα ήθελε να σχολιάσει. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου συνεισφέρει και συμβάλλει πλέον σε μια τόσο σημαντική υπόθεση όσο η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής περιοχής δικαίου, δικαιοσύνης. Τώρα στα πλαίσια των διαδικασιών αστικού δικαίου σε σχέση και με αυτά που είχαν γίνει πριν από 5 με 6 χρόνια στα πλαίσια του ποινικού δικαίου για ελάχιστα κοινά πρότυπα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων κτλ. γλωσσικά και άλλα. Ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετική είναι η κατηγορουμενων λοιπά, γλωσσικα και αλλα ηθελα να ρωτησω ποσο διαφορετικη ειναι η προσπαθεια για τα ελάχιστα κοινά πρότυπα της ε, διαδικασίας του αστικού δικαίου. Τώρα το διακύβευμα, ο στόχος, είναι το παράγωγο δίκαιο ή εν το soft law. Αλλά σήμερα το πρωί είχαμε και μία παρουσίαση από την Ιστονική Προεδρία του δικού της προγράμματος σχετικά με τις αρμοδιότητες και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ο Πρόεδρος Σλόμποντα είχε παρακολουθήσει και μία παρουσίαση του εστονικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σχετικά δηλαδή με τη συμβολή των συστημάτων του διαδικτύου. Εσείς θεωρείτε ότι θα ήταν κατάλληλο να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ευχαριστούμε την κυρία Χαούταλα. Κάποιος άλλος που θα επιθυμούσε να σχολιάσει, αν όχι, παρακαλώ, δίνω το λόγο στους ομιλητές για να απαντήσουν. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, λέει η κυρία Βόλι είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνει κανείς με το ποινικό δίκαιο. Πρώτον διότι υπάρχει τεράστιο επίπεδο δραστηριότητας ε, σε επίπεδο δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αστικό και εμπορικό πεδίο ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε με το ποινικό δίκαιο και κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί ότι τότε αυτό θα σήμαινε ότι θα ήταν πιο εύκολο Παράλληλα όμως είναι και πιο περίπλοκο διότι και είμαι βέβαιη ότι η Κομισιόν θα συμφωνεί ο Ευρωπαίος Νομοθέτης έχει αγγίξει διάφορες μικρές περιοχές της αστικής δικονομίας και διαδικασίας με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως συνολικά, όπως συνήθως ακούμε, υπάρχει μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση, μια έλλειψη συνέπειας σε βάση περιπτώσει. Και αυτό επιχειρούμε τώρα να κάνουμε στα πλαίσια του αστικού δικαίου, όχι μόνο για να αποτυπώσουμε το που βρισκόμαστε, αλλά και για να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις και δυνατότητες για το μέλλον είμαι σίγουρη ότι και η συνάδελφος θα μπορέσει να πει πολλά περισσότερα για το e-justice, αλλά οπωσδήποτε συνεργαζόμαστε και με τους αρμοδίους σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και του Ινστιτούτου και στο μέτρο του δυνατού επιμένουμε ότι αυτό το μέσο Παράγου δικαίου θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για να το πούμε έτσι για το μέλλον ένα αντιμελλοντικών αναθεωρήσεων δηλαδή. Πάντως θεωρώ ότι όπως είπε και η Εύα αργά και σταδιακά σε μια νέα τεχνολογική εποχή οπωσδήποτε κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε αυτές οι διαδικασίες να συνδυάζονται κατά κάποιον τρόπο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Όπως και η περιοχή στην οποία τίθεται. Διότι ερευνώντας ως νομικός τα θέματα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, πολύ γρήγορα πέφτει πάνω στα τεχνικά ζητήματα. Το εστονικό παράδειγμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το έχουμε εξετάσει και στην ομάδα και αυτό που είπαμε στα υπηρεσιακά έγγραφα είναι ότι για να λειτουργούν οι ίδιοι κανόνες και εθνικά και διασυνοριακά πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή πρόσβαση μεταξύ συστημάτων. Δηλαδή εγώ ως δικαστικός λειτουργός ή ως νομικός εκπρόσωπος θα έπρεπε να μπορώ μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου να επικοινωνώ με κάποιον στην Εστονία όχι αναγκαστικά σε μια ενοποιημένη διαδικτυακή πύλη, δεν τολμήσαμε καν να προτείνουμε κάτι τέτοιο, αλλά για να χρησιμοποιεί κανείς τους ίδιους κανόνες πρέπει να έχει πρόσβαση στα ίδια ηλεκτρονικά συστήματα. Τεχνικώς βεβαίως δεν έχουμε παράσχει μια τέτοια λύση και επαναλαμβάνω δεν έχουμε τολμήσει να προτείνουμε μια πλατφόρμα για όλη την Ευρώπη αλλά θεωρούμε ότι θα ήταν πιο εύκολο στο βαθμό που κατανοώ και εγώ τη δουλειά που γίνεται σε επίπεδο e-justice και από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο αυτό μια κατανεμημένη πρόσβαση θα ήταν ένας καλύτερος τοπικός τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα. Mr. Rosner, yes, if you want to add something. Thank you. Thank you for this uh, um, indeed. Ο κύριος Ρόσνερ, ευχαριστώ και εγώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ε, σχετικά με τις διαφορές ποινικού και αστικού δικαίου, όπως είπε και η κυρία Wallace το 68 ξεκινήσαμε στα του ποινικού. Από την πρώτη σύμβαση Βρυξελών και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, της ε, τους δικονομικούς κανόνες, μέχρι το Βρυξέλλες 2α για τα οικογενειακά, μέχρι καθαρά ευρωπαϊκές διαδικασίες. Έχουμε τέσσερα μέσα την εντολή ε, την εντολή για τις πληρωμές, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και στοιχεία. Ε, έχουμε ένα σημαντικό αριθμό κεκτημένου αλλά και ποιότητα κεκτημένου στο πεδίο αυτό. Και ήταν μάλλον ευκολότερο να αναπτύξει κανείς ένα κεκτημένο σε μια παρθένα περιοχή σε σχέση με τη ζούγκλα ή εμπασχετός το πλουσιότατο δάσος που είναι το αστικό δίκαιο. Για τις οδηγίες νομίζω η Επίτροπος το ανέφερε την περασμένη εβδομάδα και δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε αλλά απλώς θα πω ότι αυτή τη στιγμή εξετάζει η Κομισιόν τους καλύτερους τρόπους να προχωρήσει, διαφορετικές πηγές από των οποίων θα βασιστεί το Έλλη Ουνιντρούα για να προχωρήσει. Βέβαια είναι μια δυναμική διαδικασία εν εξελίξη. Και για το e-justice Αυτό είναι ένα έργο που κυρίως αφορά στη συνεργασία των κρατών μελών και έχουμε και έναν συνάδελφο από την ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνη που γνωρίζει περισσότερα και θα μπορούσε και να προσθέσει αλλά μία από τις περιοχές που μπορούν να εξεταστούν είναι ακριβώς το θέμα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών uh, της ηλεκτρονικής επιδόσεως εγγράφων μέσω εφισταμένων εθνικών συστημάτων ή και χωριστής πλατφόρμας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα μπορούσε να τολμήσει κανείς να πει Υπάρχουν όμως διάφορες διασυνδεδεμένες πτυχές και η Εστονική Προεδρία θα ήθελε να εξακολουθήσει να κοιτάζει το υφιστάμενο έργο που εξετάζει το e-Codex που είναι οι τεχνικές τράπεζες δεδομένων. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Προεδρεύουσα κυρία Φεράρα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ενδιαφέρουσα ακρόαση. Και να προχωρήσουμε τώρα. Ή μάλλον να επιστρέψουμε στο 14 για να μπορέσει η κυρία Γκούταλα να κάνει μια σύντομη ε, παρατήρηση για την έκθεση για την για τις αποζημιώσεις για περιβαλλοντικές ζημίες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και εσάς και τη Γραμματεία που μου επιτρέπει να τοποθετηθώ, διότι το θέμα αυτό άλλαξε ε, ε, τη σειρά του στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ και την Λάουρα Φεράρα για το έργο της, ε, που έχει σημασία. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να σχολιάσω την δική μου τροπολογία, μάλλον δύο τροπολογίες, 16 και 45, ώστε να περιληφθεί και η ατμοσφαιρική ρήπανση από καυσαέρια αυτοκινήτων. Όπως έχουμε ξαναπεί παλαιότερα, ο ορισμός του κατοφλίου για την ζημία ώστε να θεωρηθεί αυτή η πλέον περιβαλλοντική είναι πολύ υψηλό. Γι' αυτό πρότεινα τροπολογία για να θέσω το θέμα. Θεωρώ ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες πλέον για την ατμοσφαιρική ρήπανση εφόσον θέλουμε να ισχύει η αρχή ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Γι' αυτό και θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αποζημίωσης για ζημίες στην ανθρώπινη υγεία που προέρχεται από ρήπανση, που προέρχεται από αυτοκίνητα. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο πρόημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της, της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, η οποία προκαλεί καρδιακιακές παθήσεις μεταξύ άλλων. Όπως γνωρίζουμε, χάρη στις επιστημονικές έρευνες, η ατμοσφαιρική ρήπανση που προέρχεται από ε, τη βιομηχανική ρήπανση αλλά και από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλοντος ε, γενικότερα. Χρειάζεται λοιπόν να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή ώστε να περιλάβει και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καλέσουμε έντονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 32, πιστεύω ότι χρειάζεται να θεσπιστούν μηχανισμοί συλλογικής αποζημίωσης για όλα τα άτομα και οργανώσεις που έχουν υποστεί ζημίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τι δυνατότητε για θέσπιση ενό μηχανισμού συλλογική αποζημιώσεω για ζητήματα υγεία που προέρχονται από την ε, ρήπανση, από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Τα είδαμε αυτά και με την υπόθεση Volkswagen, όπου οι Ηνωμένες, ή μάλλον στι Ηνωμένε Πολιτείε η εταιρεία αυτή αντιμετώπισε συλλογικές συλλογικέ αγωγέ από καταναλωτές, από οργανώσεις αλλά και από ε, κυβερνητικές αρχές. Με την συλλογική αυτή ε, δράση μπορεί η αποζημίωση να είναι πιο αποτελεσματική. Δεν λέω ότι θα χρειαστεί να μεταφέρουμε ακριβώς το ίδιο σύστημα όπως αυτό που ισχύει στις ΗΠΑ εδώ στην Ευρώπη, αλλά ο μηχανισμός συλλογικής αποζημίωσης διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των που έχουν υποστεί ζημία από την ε, ρήπανση. Είναι σωστό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα να εξετάσουν τις σχετικές δυνατότητες. Οι συλλογικές αποζημιώσεις θα είναι αναγκαίες διότι το σύστημα αυτό θα επιτρέψει στα θύματα να ε, προβούν σε συλλογικές αγωγές, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεμονωμένα ατομικά λόγω κόστους και λόγω ε, σημαντικής ανάλωσης χρόνου. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ και πάλι την ε, γραμματεία και βεβαίω εννοώ και την πρόεδρο που μου έδωσε την ευκαιρία να τοποθετηθώ και πάλι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο, την ευχαριστώ για τις τροπολογίες της, συμφωνώ μαζί της, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και τη βλάβη στη δημόσια υγεία από τις εκπομπές καυσαερίων των αυτοκινήτων οχημάτων. Είμαι υπέρ λοιπόν των τροπολογιών της και νομίζω ότι αυτού του τύπου τη ζημία θα πρέπει να την συμπεριλάβουμε και να δημιουργήσουμε και τράπεζες δημόσιες ανοιχτές δεδομένων έτσι ώστε να καταγγέλλονται αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται τις ρυθμίσεις. Τώρα θα διακόψουμε μέχρι τις 5 και 4. Grazie.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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Dear colleagues, may we start? Ας αρχίσουμε αγαπητοί φίλοι. Με το υπαριθμόν 15. Είμαι βέβαιος ότι θα θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή στο Βίκ. Να σας πω λοιπόν με την ευκαιρία ότι η αποστολή διεξήχθη στις 22 έως 24 Μαΐου τρέχοντος και στόχο είχε κυρίως θέματα αστικής δικαιοσύνης και πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που λήφθηκαν μετά από την κατάρρευση του πιστοτικού συστήματος το 2008 και τις ε, ε, αλλαγές που ακολούθησαν στο δικαιικό σύστημα με ναι, συναντήσεις μεταξύ άλλων και για την βελτιωμένη νομοθεσία. Συμμετέσχουν ο ίδιος στην αποστολή, στην οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με εκπροσώπους υψηλωτά του επίπεδου και της πολιτικής και της ε, δικαστικής ε, ζωής. Ο δε κύριος Γιωχάνεσον, ε, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και με μέλη του Αλντίγκη που είναι το Ισλανδικό Κοινοβούλιο και ανταλλάξαμε και απόψεις με νομικούς εμπειρογνώμονες εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια δύο στρογγυλών τραπεζών. Είχα μαζί μου τους κυρίους Ράντεφ, Σβιεύκα, Μαρίνιο Πίντου, την κυρία Μπερζερόν και βεβαίως και εγώ προσωπικά, Ρωτώ με αν κανείς εκ των ε, συμμετεχόντων ε, θέλει να ε, λάβει το λόγο. Εγώ κοιτάξτε θέλω να αναφερθώ στο ταξίδι αυτό που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια μικρή χώρα 330.000 ε, κατοίκων, το μέγεθος μιας μεσαίας πολιτείας στην Ευρώπη και βεβαίως είναι κράτος και έχει και το παλαιότερο κοινοβούλιο, τα παλαιότερα κοινοβούλια του κόσμου και ένα μέρος όπου ε, υπάρχει πραγματική δημοκρατία, ε, μια πραγματική ουτοπία που σημαίνει και στην διακυβέρνηση. Διαφάνεια και δημοκρατία είναι οι δύο κέρυες έννοιες που επανέρχονται στην ομιλία τους. Ε, ζουν από ε, το ψάρεμα και τον τουρισμό. Δεν έχουν βιομηχανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να σε ενδιαφέρει. Έχουν ε, και πολύ μια σχέση έντονη με, το, με, με την οικολογία. Ο τουρισμός βέβαια τους διαβρώνει. 330.000 ε, κάτι και 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Είναι πραγματικά συντριπτική η πλειοψηφία των τουριστών. Έχει ενδιαφέρον και η αντίδρασή τους στην οικονομική κρίση, την οποία επέλυσαν με δραστικό τρόπο, εθνικοποίησαν τις τράπεζες, τράπεζες έχωσαν τους τραπεζίτες στη φυλακή και του ίδιο τους πολιτικά υπεύθυνους. Στη φυλακή έχουν πολλούς στη φυλακή, αλλά ε, ε, οι υποθέσεις επιλύονται δικαστικά μέσα σε ένα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο ε, εκδίδεται η απόφαση. Ανοιχτό σοφρονιστικό σύστημα, οι άνθρωποι ζουν σε αγροκτήματα εκεί, οι κρατούμενοι δηλαδή, με την έννοια ότι ο πολίτης έστω και κατάδικος παραμένει πολίτης και μπορεί να επανέλθει να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Άρα δεν αποκλείεται απολύτω μπορεί να πάει να κάνει ψώνια ο άνθρωπο, για παράδειγμα, βεβαίως είναι νησί και παίζει και αυτό ένα ρόλο. Και η ε, φυλακή, το ε, σοφρονιστικό κατάστημα, ε, βάση περιπτώσει, έχει αυτό χαρακτήρα. Σα ευχαριστώ. Ήταν, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που μπορέσαμε να πάμε εκεί. Νίκησαν την κρίση και 7% είναι η οικονομική του ανάπτυξη τον χρόνο. Μακάρι να μπορούσε να τους μοιάσει η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν πραγματικά ε, ενθουσιάστηκα με το ταξίδι αυτό και ως ανθρωπολόγος μπορεί να διδαχθεί κανείς πολλά πράγματα. Δεν είμαι βεβαία ότι τα πράγματα που κάνουν εκεί μπορούν να προσαρμοστούν και εδώ, διότι δεν έχουμε το ίδιο ε, αίσθημα κοινότητας. Εμείς είμαστε εδώ ιδιαίτερα ατομιστές, αλλά οι ατομικιστές. Ευχαριστώ πάντως, ευχαριστώ την νομική επιτροπή που μας ευέτρεψε να πάμε στη χώρα αυτή. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά διδακτική εμπειρία. Η κυρία Πολύ χαίρομαι για τη δουλειά που κάνει η κυρία Μπιασεγό για τις φυλακές αλλά νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση το Σεπτέμβριο επ' αυτού. Τώρα, σε σχέση με την αποστολή όταν οι Ισλανδικές αρχές ήταν υπό τεράστια πίεση το 2008 για να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε με την τραπεζική κρίση. Πώς κατάφερε να παρακολουθήσει την υπόθεση η δικαστική αρχή θα πρέπει να είχαν πολύ μεγάλες υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος, offshore κτλ. Πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Μα είπαν απλώ ότι είχαν αντιδράσει αποτελεσματικά. Το ενοχλητικό είναι ότι έχουν μόνο δύο βαθμίδες, το οποίο είναι κάπως ενοχλικό για ένα νομικό Γάλλο, αν θέλετε. Υπάρχει πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ακυρωτικό, απευθείας μετά. Και ε, γνώριζαν ότι η επιβίωση της ε, χώρας περνούσε από την ε, καταδίκη των υπευθύνων. Αλλά δεν πήγαν σε λεπτομερίες που να μπορώ να σα περιγράψω σχετικά με το πώς ακριβώς έδρασαν. Προεδρο. εγώ θυμάμαι από το θέμα αυτό απλώς ότι η τραπεζική κρίση του 8 οδήγησε και σε κρίση στα κρατητήρια γιατί δεν είχαν αρκετό χώρο δεν είχαν τόσο μεγάλες φυλακές για όλους τους υπευθύνου που οδηγήθηκαν στη φυλακή. Το οποίο άπτεται αν θέλετε και της, ε, αυτής της συζήτησης που είχαμε για τις φυλακές. Τέλος πάντων με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο. Θα συνεχίσουμε in camera. Άρα θα παρακαλούσα όλους εκείνους που δεν έχουν την σχετική, εν περιπτώσει, εξουσιοδότηση να αποχωρήσουν.